διάφορες ε, επιτροπές ε, αποφάσισαν να ξεκινήσουν ε, δια... κοινοβουλευτικές διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο 69 του κανονισμού. Οι τίτλοι των πράξεων αυτών είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου και πρόκειται να δημοσιοποιηθούν στα πρακτικά της τρέχουσας συνόδου. Σύμφωνα με το άρθρο 69.4 παράγραφος 2, ορισμένοι ευρωβουλευτέ ή τουλάχιστον ο κατώτατο αριθμό ευρωβουλευτών μπορούν να ζητήσουν γραπτό μέχρι το μεσημέρι αύριο, 3η 12 Σεπτεμβρίου, να διεξαχθεί μια ψηφοφορία όσον αφορά την απόφαση αυτή για την έναρξη διαπραγματεύσεων. Αν δεν υποβληθεί κάποια αίτημα διεξαγωγή ψηφοφορία όσον αφορά την έναρξη διαπραγματεύσεων μέχρι την προθεσμία αυτή, τότε οι επιτροπέ μπορούν να ξεκινήσουν τι διαπραγματεύσει του.